πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Σας ευχαριστώ. Έχω τη χαρά να καλωσορίσω μία αντιπροσωπεία βουλευτών και άλλων επισκεπτών του Καναδικού Κοινοβουλίου και της αντιπροσωπείας του Καναδά εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πήραν θέση στο θεωρείο, το διπλωματικό θεωρείο του ημικυκλίου τα μέλη της αντιπροσωπείας είναι στις Βρυξέλλες για να συναντηθούν με τους ομολόγους τους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί τη ευκαιρία της 32ης διακοινοβουλευτικής συναντήσεως Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Καναδά. Δευτέρα και Τρίτη αυτής της εβδομάδας υπήρξε η δυνατότητα να συζητήσουν με πολλούς από τους βουλευτές μας και χθε επεσκέφθησαν την πόλη της επί τη ευκαιρία του εορτασμού ε, της ε, λήξης του Παγκοσμίου Πολέμου. Και εύχομαι καλή συνέχεια στην αντιπροσωπεία, καλή συνέχεια της διαμονής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τις επεξηγήσεις ψήφων. Επεξήγηση όσον αφορά την προγραμμάτισα των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην ευρωεκφελιστικές ασθένειες.